Λοιπόν, σύμφωνα... με την ε, απλουστευμένη διαδικασία θα πρέπει να ψηφίσουμε την έκθεση του κυρίου Κώστα για την σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη συνεργασία όσον αφορά την κανονιστική ρύθμιση της, ασφαλ... της ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας. Ονομαστική ψηφοφορία η οποία άρχεται τώρα. Le vote est ouvert. Αρχίζει η ψηφοφορία παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία για την πρώτη έκθεση του κύριου Κώστα. Tout le monde a voté. Ψηφίσατε. Πέρασε ψηφοφορίας. Υιοθετήθηκε. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη θα ψηφίσουμε με προστευμένη διαδικασία την έκθεση κυρίας Γουόλης για το κοινό καθεστώς για την εμπορία ο αλβουμίνη και γάλακτα αλβουμίνη. Ονομαστική ψηφοφορία η οποία αρχίζει. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετήθηκε. Σύμφωνα με τη μερίσια διάταξη θα ψηφίσουμε σύμφωνα με απλουστευμένη διαδικασία την έκθεση κυρίας Γουόλης για το φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μερικές διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγέ μενοχών που αφορούν εταιρείε διαφορετικών κρατών μελών καθώς για τη φορά της καταστατικής έδρας αρχίζει ψηφοφορία, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, πέρασε ψηφοφορίας. Υιοθετήθηκε και αυτή έκθεση του κυρίου Μποτόπουλου για το γλωσσικό καθεστώς που ισχύει στις αιτήσει ανέρεσης κατά των αποφάσεων του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ονομαστική ψηφοφορία η οποία ξεκινάει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας υιοθετήθηκε. Έκθεση του κυρίου Μπέλτερ για τις οικονομικές ε, και εμπορικές σχέσεις με τα Δυτικά Βαλκάνια. Ονομαστική ψηφοφορία η οποία άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετήθηκε. Έκθεση τη κυρία Γκίνα, της κυρίας Μαγκίνας μάλλον, για την κοινή γεωργική πολιτική και την παγκόσμια επιστηστική ασφάλεια. Ονομαστική ψηφοφορία η οποία αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετήθηκε έκθεση κυρίας Γκραμπόφσκα για τις προοπτικές ανάπτυξης του διαλόγου των πολιτών στο πλαίσιο της συνθήκης της Λισαβόνας, ονομαστική ψηφοφορία. ο κύριος Μπίσλη ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Φαίνεται ότι έχουμε πολλές ονομαστικές ψηφοφορίες που είναι λίγο περίεργο για μένα, διότι πραγματικά ε, δεν λειτουργεί το μηχάνημά μου. Λοιπόν, μέχρι στιγμή έχω ψηφίσει ναι και ψηφίζω ναι, αλλά να έρθει και ένας μηχανικός να μου το διορθώσει το μηχάνημα, σας παρακαλώ. Θα σας στείλουμε έναν τεχνικό αμέσως, αλλά μήπω να βρείτε